Ε, ε, Συνεχίζουμε, αφού έχουμε ολοκληρώσει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βάση της ημερησίας διάταξης θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την δέσμη μέτρων για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Uh, Παρακαλώ Νόμιζα ότι θα υπήρχε και μια διαδικασία catch the eye για τη συζήτηση αυτή, κυρία Πρόεδρε. Θα υπάρξει διαδικασία catch the eye για την δήλωση για το πακέτο χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Πρέπει να είμαι σαφής ωστόσο προς τους συναδέλφους. Δεν θα Φυστώ δευτερολέπτου στο χρόνο ομιλίας. Έχουμε πολλούς ομιλητές και μακρό χρόνο ψηφοφοριών. Όταν λοιπόν λίγη ο χρόνο σας θα σας, βγα... αφαιρώ το λόγο. Σε ό,τι αφορά το catch the eye θα πρέπει να τηρηθεί το πεντάλεπτο συνολικά. Λυπάμαι αλλά έτσι έχει σήμερα το πρωί. Δίδω αμέσω το λόγο στο Συμβούλιο. Ο κύριος Ρεντέρς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά επανέρχομαι ενώπιον σας για να ασχοληθώ και πάλι με το θέμα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας διότι είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και μετά την τελευταία συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ. Το νομοθετικό πακέτο για την εποπτεία έχει πλέον υποβληθεί στο Κοινοβούλιο προς ψηφοφορία. Πρόκειται για μια σειρά κειμένων που θεσπίζουν μια πολύ σημαντική μεταρρυθμίση στην Ένωση, ανταποκρινόμενα σε πολλέ προκλήσει. Η πρώτη είναι αυτή που σχολίασε και ο πρόεδρο του Συμβουλίου, η απάντηση στην κρίση. Στην ε, δεκαετία που λύγει, δεδομένης και της αρχιτεκτονικής λαμφαλουσή όπως ξεκίνησε, σε, όλες τις, σε όλο το πλαίσιο ε, έχουν οι επόπτες τα πρώτα τους όπλα. Αυτό συνέβαλε στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ε, οικονομικής νομοθεσίας και μια προοδευτική πολιτική ε, προληπτικής εποπτείας σημαντική και θετική για να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Βάσει της κρίσης, ωστόσο, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ολίγων φιλόδοξη. Δεν πρόλαβε, ούτε περιόρισε την οικονομική χρήση, δεν μπόρεσε να, δώσει, να συντονίσει τις απαντήσεις επιτόπου και δεν επέτρεψε μια σωστή διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστημικών, Συστημικών που συστημικών κινδύνων που θα λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υπό την εποπτεία του Πρόεδρου της είναι διαθετημένη να συνεργαστεί για την υλοποίηση και εφαρμογή της Επιτροπής αυτής. Δεν είμαι, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τρισέ θα συμβάλλει όπως μπορεί με τη γνώση και την εμπειρία του και στην παρακολούθηση πιθανής ε, πιθανών συστάσεων ή προειδοποιήσεων υπό την Προεδρία του. Για τον ίδιο στόχο θέλουμε οι να έχουμε ισχυρότερε και πιο αντιδραστικέ εποπτικέ αρχέ, έτοιμε να προετοιμάσουν κοινοτικού κανόνε και να επαγρυπνούν στην πλήρη υλοποίησή του συμπεριλαμβανομένων και των περίοδων κρίσεω. Οι αρχέ αυτέ θα έχουν τα νομικά μέσα για να επιβάλλουν το σεβασμό των κανόνων στα τραπεζικά ιδρύματα σε περίπτωση ε, αδυναμίας κάποια εθνικής εποπτική αρχής. Θα συμβάλλουν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και χώρο εποπτεία που είναι αναγκαίο για την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά. Επίση, θα συνδέονται με τη λειτουργία του, του Κολεγίου των Εποπτικών Αρχών και θα επιλύουν πιθανέ διαφορέ μεταξύ εθνικών αρχών. Ε, ε Αφήνοντα βεβαίω τι τελευταίε την διεξαγωγή τη προληπτική εποπτεία σε καθημερινή βάση. Δεν πρέπει να, να φοβόμαστε τα λόγια. Η δημιουργία των αρχών αυτών είναι μια ιστορική συμφωνία. Το είπαν ήδη ορισμένοι στο σώμα σα πολλέ φορέ η Βελγική Προεδρία θεώρησε ότι κάτι τέτοιο ήταν από τις κύριε προτεραιότητέ της στον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και συνολικά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπαίνουμε, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα πρωτότυπο μοντέλο εποπτείας, θα επανέλθω σε αυτό. Ταυτόχρονα ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη την εξέλιξη των δομών εποπτείας στου κύριου εταίρους μα. Αυτή είναι η δεύτερη πρόκληση. Να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι ικανή να μεταρρυθμίζει τις εποπτικές ε, δομές της χωρίς να απομακρύνεται ιδίω από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Με την έκθεση Ντελαροζιέρ του Φεβρουαρίου του 2009 που υποδέχθηκε πολύ ευνοϊκά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η συζήτηση στην Ευρώπη πήρε ε, σωστό δρόμο και οδηγεί στις ελπίδες μεταρρύθμισης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εντωμεταξύ ξεκίνησαν μια σημαντική αναθεώρηση των εποπτικών δομών τους με, με την υιοθέτηση του Dodd-Frank Act, ε, ψηφίζοντας σήμερα το νομοθετικό αυτό πακέτο όπως ελπίζω, καρπό ενός έτους συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναπαύεται, δεν είναι πίσω, αλλά είναι, έχει ηγετική θέση στις μεταρρυθμίσεις μέσα στο πλαίσιο των, ε, της των 20. Θα πρέπει πέραν της ε, σημερινής ψήφου ωστόσο να δείξουμε ότι εξελίσσεται το πλαίσιο αυτό. Αυτή είναι η τρίτη μας πρόκληση. Αυτό που θέλουμε είναι ένα μοντέλο μικροπροληπτικής εποπτείας, ε, ε, εκτεταμένα αποκεντρωμένο, όπου οι εθνικές αρχές οι ευρωπαϊκέ αρχέ θα συντονίζουν και θα αντικαθιστούν τι εθνικέ αρχέ. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να ενισχύεται και όχι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινδύνου δημιουργούμε ένα ουσιαστικό εργαλείο συζήτησης και λήψη αποφάσεων σε μακροοικονομικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένο και σε διατλαντικό και παγκόσμιο πλάνο. Με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα έχουμε αποτελεσματικούς δρόντες στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων εάν τους δώσουμε τις δυνατότητες ανάληψης δράσεων. Αυτό συμβαίνει με την οδηγία Omnibus 1 που, επί του οποίου θα λάβει θέση το Κοινοβούλιο σήμερα. Στα, τα, τα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ωστόσο, έχουν επίσης σημασία και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε και κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές να σταματήσω εδώ. Φτάνουμε σήμερα στο τέρμα μιας πρώτης κρίσιμης φάσης. Ελπίζω ότι η ψηφοφορία αμέσως μετά θα είναι θετική. Θέλω ωστόσο να ευχαριστήσω την, ιδιαίτερα τους, ε, τον την πρόεδρο της ε, Επιτροπής, τους διάφορους ε, εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και τον Επίτροπο Ρεν και τον Μισελ Μπαρνιέ παρόντες εδώ, αλλά και όλους τους συνεργάτες τους. Είχαμε με όλους αυτούς καρποφόρες και προφανώς επικοδομητικές ανταλλαγές που επέτρεψαν να υποβάλλουμε σήμερα αυτό το τροποποιημένο κείμενο. Θα ήθελα η βούληση ε, ολοκλήρωσης που μας ενέπνευσε ναι, ναι, να συνεχίσει να συμβάλλει και στις επόμενες διαπραγματεύσεις για τα προσεχή κείμενα που θα ανανεώσουν και θα ενημερώσουν το θεσμικό πλαίσιο. Δεν θέλω να δεσμεύσω τους διαδόχους μου στους, στην Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά βάσει των τελευταίων διαπραγματεύσεων είμαι βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί και ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα επανέλθουμε με νέε συμφωνίε, ιδίω στον τομέα, τομέα των επενδυτικών ταμείων, μαζί με τον Επίτροπο κ. Μπαρνιέ να υποστηρίξουμε ένα πλήρε χρονοδράγμα δράσεων για την υλοποίηση του νέου αυτού νέων νομοθετικών κειμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η συμφωνία επί της οποίας θα εκφράσετε γνώμη τόσο λίγο που αφορά τις, ε, τις διατάξεις της εποπτείας προέρχονται από μια πρόταση της Κομισιόν και μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα στην εξέλιξη της, ε, της χρηματοοικονομικής ρύθμισης της Υπήρου μας αντέδρασε η Κομισιόν στην διεθνή κατάσταση, εισήγαγε στη διαδικασία των G20 στη διάσκεψη της Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2008. Η ομάδα εργασίας ε, κατέληξε στα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση και ευθύς εξ αρχής η Κομισιόν διατύπωσε τις ε, προτάσεις της. Θέλω να αποτίσω, να τιμήσω την ευφυή εργασία του Ζακ Ντολαγουζιέ, στον οποίο οφείλουμε πολλά. Με αυτή τη συμφωνία διαθέτουμε, αν θέλετε, ένα πλαίσιο εντός του οποίου πλέον θα κινούνται όλες οι πρωτοβουλίες που προϊόν προς προϊόν, αγορά προς αγορά, από οικονομικό παράγοντα προς οικονομικό παράγοντα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε. Στις 13 Ιανουαρίου του 2010, κατά την ε, ακρόασή μου, μία λοιπόν αποτελεσματική διοίκηση. Αυτό το πλαίσιο το οποίο εγκρίναμε αποτελεί τη βάση που καθιστά αξιόπιστες όλες τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε σε κάθε τομέα. Η συμφωνία αυτή οφείλεται στην προσωπική δέσμευση και την γνώση πολλών από εσά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές Monsieur Καθώς και το σκιώδη εισηγητή την Sharon, Bowles που ξεκίνησε αυτή τη διαπραγμάτευση με πολλή αποφασιστικότητα. Επίσης, Didier Hinders τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ για την προσπάθεια που έκανε αυτός και οι συνεργάτες του που ήταν καθοριστική για να στηριχθούμε στην καλή δουλειά που έκανε πριν από αυτόν η Ισπανική και η Σουηδική Προεδρία. Και θα ήθελα κατά τρόπο αρκετά ασυνήθιστο να σας, και θα σας εξηγήσω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους Κομισιόν αυτόν που βρίσκεται εδώ δίπλα μου, τον David Wright γιατί θα φύγει από την ε, θέση του που είναι βοηθός Γενικού Διευθυντή για τις ε, χρηματοοικονομικές υποθέσεις. Πρέπει να πω αυτό που σκέφτομαι. Ο άνθρωπος αυτός αποτεί τιμή στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Αποτελεί τιμή για μας. Η προστιθέμενη αξία, κυρίες και κύριοι, του Κοινοβουλίου αποτελεί ένα σταθερό και καθοριστικό παράγοντα και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ε, ε, εποπτικής αρχής, την διαμεσολάβηση των κατεπηγόντων, την προετοιμασία των τεχνικών και νομικών διατάξεων, την πρόληψη και την προστασία από κάποια τοξικά προϊόντα το διαμεθοριακό εμπόριο και βεβαίως και θέλω να ευχαριστήσω τον Όλη Ρέν, τον συνάδελφο και τους συνεργάτες του που δημιούργησαν αυτό το που αφορά τους συστημικούς κινδύνους. Βεβαίως όλα αυτά θα αποτελέσουν συμβιβαστική πρόταση. Άλλοι θέλαν να προχωρήσουν περισσότερο. Η Κομισιόν σε πολλά θέματα έκανε δυναμικές, δυναμικούς συμβιβασμούς, παραχωρήσεις. Έχουμε ας πούμε την διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προτύπων που δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για άλλους τομείς, θέλω να το δηλώσω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει συνολικά η ψήφος του Συμβουλίου, με τη δική σας ψήφο σήμερα αν το θελήσετε, θα μπορέσει να χαρίσει στην Ευρώπη από την αρχή του επόμενου έτους ένα μοντέλο εποπτείας ανάλογο με τις ανάγκες της, ανάλογο με τις ε, ανάγκες που έχουν οι τράπεζες που ανήκουν στις χώρες μας. Αυτή είναι η διεθνική διάσταση και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και των κινδύνων που μπορούν να αναλάβουν. Έχουμε λοιπόν μια εποπτεία κατάλληλη που θα μας επιτρέψει να, προκαταλάβουμε τις ε, κρίσεις. Ε, οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι η Ευρώπη αντέδρασε, ότι έμαθε από την κρίση και ότι προχωρούμε παράλληλα με τους Αμερικανούς και ίσως και με άλλες υπήρους για το στο πλαίσιο των G20. Όσον αφορά τις αρχές και για να υπάρξουν τελικά και να είναι αποτελεσματικές από την 1η 2011 έχω ενώπιόν μου, εγώ δηλαδή, να κάνω μια πολύ σημαντική δουλειά δημοσιονομική και τεχνική. Με την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου θα ορίσω τον Πρόεδρο και τους Γενικούς Διευθυντές αυτών των αρχών και θα σας πω ότι το μοναδικό κριτήριο που θα διέπει αυτούς τους ε, διορισμούς θα είναι η ανεξαρτησία και η δυνατότητα να οδηγήσουν στις αρχές αυτές σε επιτυχία. Όπως είμαι πεπισμένος ότι ο, ο επόμενος πρόεδρος ε, της επόμενης αρχής συστημικού κινδύνου θα έχει τις ίδιες δυνατότητες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε για να, γεμίσουμε αυτό το πίνακα που θα έχουμε ενώπιόν μας από την 1η Πρώτου 2011. Χάρη στο ρόλο που θα έχουμε από, τον, ε, από τις αποφάσεις που έχουν ή που θα ληφθούν. Θα έχουμε ε, σχέδια κανονισμών για τα παράγωγα και για τα credit fault swaps, τα οποία ήδη έχουν ε, διεκπαιρεωθεί. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να εξηγιάνουμε, για να κάνουμε διαφανέστερο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, βήμα προς βήμα δίπλα σας, μαζί σας μια σειρά από θέματα από τον οποίο δουλεύουμε θα συμφωνήσουμε, ε, ε, θα υλοποιήσουμε την Βασιλεία 3 η οδηγία για τις χρηματοοικονομικές αγορές, ενίσχυση των κυρώσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της οδηγίας για την αγορά, η δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κρίσεων. Όλα αυτά τα μέτρα θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε την επανάληψη σοβαρών κρίσεων, θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές που είναι και φορολογούμενοι και να ε, ενδυναμώσουμε την δίκαιη ανάπτυξη που θέλουμε να πετύχουμε. Κυρίες και κύριοι, και στον τομέα των χρηματοοικονομικών και στο περιβάλλον η πρόληψη είναι πολύ φθηνότερη από την ε, διόρθωση. Πρέπει με τον α ή β τρόπο να κινητοποιήσουμε το 17% για το, του ΑΕΠ ε, της Ευρώπης για τη διάσωση ε, του, της ε, ε, οικονομίας από την κρίση. Οι τράπεζες θα πρέπει να πληρώσουν για τις τράπεζες. Αυτά είναι τα μέτρα που θα υποβάλουμε στο πλαίσιο της ατζέντα που ενέκρινε η Κομισιόν και στήριξε το Συμβούλιο Κοφίν τις 2 του περασμένου Ιουνίου. Έχουν υλοποιηθεί και παρουσιάζονται με αποφασιστικότητα. Ψηφίστε τα αν θέλετε για να, να, μπορέσει να τα παρουσιάσει η ε, Κομισιόν πριν το τέλος του 2011. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προσωπικά θέλω να πω η ποιότητα των σχέσεών μας, η εμπιστοσύνη μας που δεν βεβαίως συνεπάγεται και κάποια ε, χαλαρότητα, ε, δείχνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχουν οι αγορητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ξεκινώ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κ. Γκαρσία Μαγκάγιο. Για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μια καλή μέρα σήμερα για την Ευρώπη. Το Δεκέμβριο είχαμε μια κακή συμφωνία και σήμερα χάρη στη συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, τη Προεδρία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έχουμε μια καλή συμφωνία πλέον. Μια καλή συμφωνία που θα καθορίζει αρχές που θα είναι αυθεντικά ευρωπαϊκές, αρχές ισχυρές και αρχές που θα υπόκεινται στον δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο από την Ευρωβουλή. Αρχές που θα επομιστούν και θα επιφορτιστούν και θα σχεδιαστούν ώστε να διασφαλίζουν ότι όλες οι τράπεζες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και κανονισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την επιβολή των αποφάσεων στους επιτηρητές Εθνικού επιτήρητέ, σε περίπτωση που ε, δεν υλοποιούνται οι στόχοι όσον αφορά τι ε, ιδιωτικές τράπεζες. Προστασία στι οικογένειε και στις επιχειρήσει, Ανακούφιση στι τράπεζε που μπορούν να προκαλέσουν συστημικού κινδύνους. Και θα αποφύγουμε έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να ξαναπληρώσουν, να πρέπει να ξαναπληρώσουν για τις αλόγιστε δράσει ε, θεσμικών οργάνων. Το μάθημα από αυτή τη συζήτηση ποιο είναι. Είναι ότι αυτή η Ευρωβουλή δεν είναι ένα σκυλί που γαυγίζει και υποχωρεί όμως και βάζει την ουρά κάτω από τα σκέλια όταν ε, του επιβάλλει κάτι το Συμβούλιο ούτε είναι ένα σκυλί το οποίο ούτε τρώει ούτε αφήνει άλλους να φάνε. Είναι ένας καλός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για να προχωρήσουμε θετικά στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ τους κοινοβουλευτικούς συναδέφους, τους εισηγητές, τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τον Υπουργό Ρέντερς. Έχουμε σήμερα μια εξαιρετική συμφωνία και έτσι λοιπόν μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας. Ο κύριος Κίν, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον ε, Επίτροπο, τον κύριο Ρέιντερς και τον David Wright. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα. Ε, είχαμε μια επιτυχία, αλλά ή σε παρασύρει στιγμή ή την παρασύρει. Η χρηματοοικονομική κρίση έχει δημιουργήσει νέους οργανισμούς χρήσιμους και ευπρόσδεκτους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή δημιουργησει νεους οργανισμους χρησιμου και ίσως και στον ολόκληρο τον κόσμο. Η εξουσία που θα δοθεί σε αυτούς τους θεσμικούς οργανισμούς πρέπει να είναι μια σοβαρή εξουσία. Πρέπει να υπάρχει φιλοδοξία και να υπάρχει σκοπιμότητα η σκοπιμότητα αυτή πρέπει να, γίνει αντιληπτή και από τους πολίτες που εξαρτώνται από εμά. Η συζήτηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο έχει οδηγήσει σε εντάσεις συχνά. Αλλά κανένας μας δεν πέτυχε όλα όσα ήθελε, ενώ ταυτόχρονα όλοι καταφέραμε να πετύχουμε, μια... να οδηγήσουμε σε μια επιτυχία. Έχουμε ε, περισσότερες εξουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση φυσικά και ε, την κατάσταση στα κράτη-μέλη και παρά την επιθυμία τους. Κάποιοι εδώ θέλαν να προχωρήσουν περισσότερο, να υπάρχει απευθείας εποπτεία. Ε, και όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για μια περιπετειώδη, φιλοδοξία. περιπετειώδους φιλοδοξίας. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε κάποια κενά αργότερα. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα τώρα στηρίζεται σε εμπειρία δεκατιών από ανθρώπους που έχουν εμπειρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και οι εθνικές κυβερνήσεις έδειξαν ότι μπορούν να μας σώσουν στην περίπτωση καταστροφής. Αλλά αυτό ήταν μοιραίο, δεν ήταν σχεδιασμένο. Θα πρέπει αυτά τα θεσμικά όργανα να μας δώσουν ένα σχέδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν ο σκοπός τους να εκπληρωθεί. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πρακτικά θέματα υπάρχει μια κοινή επιτροπή που με χαρά προώθησε αυτά τα θέματα. Πρέπει να αποτελέσει μέσο συντονισμού ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή λήψη αποφάσεων. Θα αποτελέσει τη βάση για να στραφεί η δουλειά αυτών των οργανισμών για, να εντοπιστούν η συστημική κίνδυση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παρακολουθεί τον κίνδυνο, αλλά αν πρέπει να ρωτήσουμε ο κύριος Μπερνάκη αν βελτιώθηκε η φήμη του, νομίζω θα πει όχι παρά τις εξουσίες. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τις πολιτικές τύπου καζίνου του παρελθόντος και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε ως ρυθμιστικές αρχές μετρημένα. Βεβαίως οι φιλοδοξίες στηρίζουν τις ε, οικονομίες και τις συντάξεις των ανθρώπων. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η επιτήρηση, είναι νέα αλλά θα πρέπει να μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Σκίνερ, δέχεστε μία ερώτηση από τον κύριο Ντάτμορ. Παρακαλώ. Με ποια βάση θεωρείτε, πάνω σε ποια βάση θεωρείτε ότι η κρίση και οι αποφάσεις νέων ευρωπαϊκών οργάνων θα είναι καλύτερες από αποφάσεις που λαμβάνουν τα εθνικά, ή εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αν είχατε ακούσει αυτά που έλεγα, θα το καταλαβαίνετε. Είπα, χρειάζεται συντονισμό με τι εθνικέ αρχέ, όχι ει βάρο των συμφερόντων του και να γίνεται μόνο όταν η νομοθεσία που προωθούμε για το σκοπό αυτό έχει εγκριθεί βάσει των δημοκρατικών διαδικασιών στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό καλύπτει το καλύτερο και των δύο πλευρών. Εάν επιμένετε να μένετε σε ένα νησάκι μόνοι σα και πιστεύοντα ότι θα προστατευτείτε έτσι από τους κινδύνους του πραγματικού κόσμου, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Ο κόσμος και η σημερινή οικονομική κρίση μας έδειξαν το μάθημά μας. Ευχαριστώ για του φιλελεύθερου. Η κυρία Μπόλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε προεδρεύων. Πετύχαμε. Η εποπτική αρχιτεκτονική μπήκε στο τρένο και ξεκίνησε φεύγοντας από το σταθμό. Ελπίζουμε ότι θα δώσει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, η οικονομική νομοθεσία ε, παραμένει ακόμα σαν ένα ελβετικό τυρί. Έχει πολλά, πολλές τρύπες, πολλά κενά σημεία όπου η ενιαία προσέγγιση δεν θα φτάσει ποτέ. Και αυτό είναι κρίμα, ένα κρίμα για όλους μας που θα παραμείνει έτσι μέχρι ότου πραγματικά τηρήσουμε την ενιαία αγορά στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι νέες αρχές μας δίνουν μια νέα διάσταση για να επιτύχουμε συντονισμό σε διασυνοριακό επίπεδο. Τούτο ωστόσο απαιτεί να, να προσέξουμε καλύτερα για να μπορούν οι αποφάσεις μας να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι κοντά στην αγορά. Η Ένωση θα πρέπει να ε, η ευρωπαϊκή προσέγγιση θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές και πραγματικά για να αποφασίσουμε πρέπει να υπάρχει ο συντονισμός όλων. Η καλύτερη απόφαση βεβαίως κατά ανάγκη είναι αυτή που είναι πιο ε, διευρυμένη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Γκίγκολτ, δύο λεπτά. Ε, Σήμερα βάζουμε ένα επιπλέον λιθαράκι στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού μας σπιτιού. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέγαμε ότι θα ξεκινήσει μια φάση επανεθνικοποίηση σε αυτή τη φάση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Ευρώπη καταλήγει σε συμπεράσματα με βάση τη συνέβη, αλλά βεβαίω πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την νομοθεσία που αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Έχουμε καταφέρει με νομοθετήματα, με την συνεργασία όλων των δυνάμεων στο σώμα και έτσι αντισταθήκαμε στους πειρασμούς κάποιων κρατών μελών να μην συναγάγουν συμπεράσματα από αυτήν την κρίση. Παραμένουν κάποια σημαντικά θέματα εκκρεμή. Για παράδειγμα το θέμα ποιο θα είναι το προσωπικό, πόσα άτομα θα έχουν αυτές οι υπηρεσίες. Τι χρησιμεύει να υπάρχουν νέες υπηρεσίες αν δεν υπάρχουν τα αναγκαία στελέχη Έχουμε κάποια μηνύματα ότι δεν είναι σαφή αυτά τα πράγματα. Θα καταβάλουμε προσπάθειες να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Επόμενο ερώτημα. Τι θα γίνει, α το πω έτσι, με τον πρόεδρο αυτών των αρχών, χρηματοοικονομικών αρχών. Και εκεί θα μεριμνήσουμε να επιλεγούν οι σωστοί άνθρωποι. Για μας ως Πασίνου, ήταν σημαντικό βήμα επιτέλου να υπάρξει διαφάνεια. Αυτό θέλαμε μέσω και των διαφορετικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις πολυεθνικές να υπάρξει διαφάνεια. Τώρα χαιρόμαστε ότι προανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για το country by country reporting την σύνταξη εκθέσεων ανά χώρα θα υπάρξουν εκθέσεις. Χαιρόμαστε για το κοινό έργο που πρέπει να επιτελέσουμε. Υπάρχει και στο τέλος μια κοινή δήλωση των τεσσάρων συντονιστών στην ΕΚΟΝ, στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων, ότι θέλουμε να εμπλακούμε και να ε, δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τη στελέχωση. Μια τελευταία παρατήρηση. Ελπίζω ότι στο θέμα της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης θα υπάρξει η ίδια συνάφεια και συνοχή από το σώμα όπως και στο παρελθόν. Γιατί διαφορετικά δεν θα ασκήσει την επιρροή του το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν πρέπει να κατακαιρματίσουμε τη συζήτηση. Κατά τα άλλα, δυστυχώς το Συμβούλιο δεν θα αποφασίσει σωστά πράγματα αν εμείς δεν δράσουμε όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για τους ε, Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές και συντηρητικού, ο κύριος Σουίλμπορν, δύο λεπτά. Η κυρία Σουίλμπορν, η κρίση δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας στον οικονομικό τομέα. Οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις το αισθάνονται αυτό σε καθημερινή βάση και οι οικονομολόγοι λένε ότι για να υπάρξει ανάκαμψη θα πρέπει αυτή η αβεβαιότητα να πάψει να υπάρχει. Ένα από τα βασικά προβλήματα της τεράστιας αποτυχίας στον τομέα ήταν η εποπτεία, μεταξύ των οποίων και ποιος θα κάνει την επερχόμενη εποπτεία. Ε, το σώμα μας, το Κοινοβούλιο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σχετική συζήτηση για το ποιος, πότε, πού και πώς θα πραγματοποιηθεί η εποπτεία. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο μεταξύ ευθυνών κρατών μελών για τα εποπτικά του ιδρύματα και μια νέας Ευρωπαϊκή αρχής ε, που θα θέτει κοινού κανόνες, προωθώντα κατά συνέπεια την ενιαία αγορά στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιτρέποντας καλύτερη εποπτεία από, τους, ε, ε, από τις ισότιμες δομές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει με ισορροπία μεταξύ κινδύνων και ασφάλειας, μεταξύ κεφαλοκρατικής και ε, προστατευτικής οικονομίας, δημιουργώντας ανεξάρτητες δομές παρακολούθησης αγοράς διαχείριση του παγκόσμιου κινδύνου από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, εξασφαλίζοντα συντονισμένη διαδικασία σε όλα τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια μια κρίση, εξασφαλίζοντα καλύτερη ρύθμιση και διαμεσολάβηση μεταξύ εποπτικών αρχών, ενισχύοντας την εφαρμογή των κανόνων από όλε τι δομέ και σε κάθε ε, σημείο. Το εποπτικό πακέτο έχει τώρα αποτελεί τη σωστή ισορροπία. Συγγνώμη, μπορείτε να μιλάτε λίγο λιγότερο γρήγορα. Ωστόσο, η πρόσληψη ε, ικανού προσωπικού θα είναι βασικό για την επιτυχία του, της διαδικασίας. Ζητώ λοιπόν να εξασφαλίσει ότι το επόμενο βήμα ε, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το επόμενο βήμα θα τηρηθεί. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Κλούτ, δύο λεπτά. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους που εδώ πέρυσι και μάλιστα σε μακρόχρονες ε, διαπραγματεύσεις είχαν εμπλακεί, να τους ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη επίδοση του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών το ότι κατάφεραν αυτό που πέτυχαν. Ήταν το βέλτιστο το οποίο μπορούσε να επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, υπό το πρίσμα της ομάδας μου, της ε, επικρίσεις που έχουμε δεν θα τις παρασιωπήσω. Κυρίως τρία σημεία είναι εκείνα τα οποία μας δυσαρεστούν. Αφενός το σημείο το ότι υπό το πρίσμα μας οι αρμοδιότητες δεν είναι επαρκείς όσον αφορά τις εποπτικές αρχές. Αυτές οι αρμοδιότητες που τους δόθηκαν θα το χαιρετίζαμε αν είχαν περισσότερες αρμοδιότητες. Το θεωρούμε ένα σφάλμα επίσης το ότι οι εποπτικές αρχές επιμερίζονται σε διαφορετικές έδρες. Είχαμε προσπαθήσει και ζητούσαμε σε μία έδρα να συγκλίνουν και να έχουν την έδρα τους όλες αυτές οι αρχές. Αυτό θα διευκόλυνε το έργο. Και προηγούμενα αναφέρθηκε κιόλας σε σχέση με τα στελέχη η στελέχωση θα έπρεπε μακροπρόθεσμα να διασφαλίζεται με καλύτερο τρόπο. Αυτές είναι οι επικρίσεις μας. Παρ' όλα αυτά το θεωρούμε σημαντικό και ορθό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για τη νέα ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών που είναι επιτακτική και επίγουσα ανάγκη. Όμως, Επίσης θέλω να δώσω την εκτίμησή μας ότι επιτέλους πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα περαιτέρω βήματα επιπλέον ώστε να καταλήξουμε σε μια πραγματική νέα εκ νέου ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών ώστε να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου Μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών και κανόνων, μια τέτοια κρίση στο μέλλον θα μπορεί να αποφευχθεί πλέον, σαν αυτή που ζήσαμε στο παρελθόν. Θα καταβάλουμε προσπάθειε ω ομάδε εμεί. Υπάρχουν κάποια νομοθετικά εγχειρήματα τα οποία βρίσκονται καθοδόν. Ελπίζουμε ότι κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αποκτήσουν σάρκα και οστά, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Αλλά πιστεύω κάποια βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ για την προσοχή για την Ευρώπη, για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ο κύριος Μπλουμ. Δυόμιση λεπτά. Κύριε Πίτρο, την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, όταν το συναντηθήκαμε δηλαδή, είχα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. Διότι θα πήγαινε η ρυθμιστική αντιμετώπιση του ΣΥΤΙ στις Βρυξέλλες και ξεπλάγεται από τις ανησυχίες μου. Έκτοτε ωστόσο μπορεί να καταλάβατε μετά την ανάληψη των ε, ευθυνών σας ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της Βρετανίας προέρχεται από τις οικονομικές υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικές για το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα καλύπτει τα κενά, τα περισσότερα κενά. 45 εκατομμύρια λίρες την ημέρα στέλνονται εδώ για να υποστηρίξουμε το ύποπτο κάπως ευρωπαϊκό εγχείρημα που χωρίς ωστόσο να δίνει στους εκλογείς μας ε, δικαίωμα λόγου. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό και πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεγάλες ε, συντάξεις, οι μεγάλοι μισθοί δεν ε, βγαίνουν, δεν, δεν κρέμονται από τα δέντρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις, ε, τα διάφορα ντομίνιον της Βρετανίας που, που ταλαιπωρούνται. Τότε μας είχατε πει έτσι με κάπως φρασί θα έλεγα τώρα, ότι μακριά είναι η Αυστραλία. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση στέκει ακόμα. Κύριε Πίτροπε, ωστόσο ακόμα και τώρα ανησυχώ ότι ε, θα υπάρξει μια ρυθμιστική προσέγγιση από τη συνηθισμένη ε, ομάδα των άσχετων ε, δημοσιονομικών υπαλλήλων της Επιτροπής που ακούνε τις απόψεις του Κοινοβουλίου που είναι κάτι οι Γερμανοί, κάτι περιθωριακή πράσινη και άλλοι. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά εγχειρήματα, την αλληλεία, τη γεωργία, την απασχόληση, τη μετανάστευση και την ορολογιακή βόμβα του ενιαίου νομίσματος. Μια εντυπωσιακή αποτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζεται ότι θα μπορέσει ποτέ κάτι να πετύχει σωστά κατά λάθο. Λυπάμαι, δεν είμαι ικανοποιημένο. Είμαι εξαιρετικά οργισμένος που οι Βρετανοί συντηρητικοί έδωσαν, παρέδωσαν την νομοθετική ρύθμιση του ΣΥΤΙ. Αν ήταν ο Τραφάλγαρο Κάμερο, το άγαλμα στην πλατεία του, στην πλατεία θα ήταν του Βιλνέβα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος... Ο κύριος Σώσα Βάγνερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Συγχαίρω εκείνους που εργάστηκαν για αυτή την έκθεση σε αυτό το πακέτο δέσμη μέτρων για τα χρηματοοικονομικά. Και επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω και τα στελέχη. Χρειάστηκε μια χρηματοοικονομική κρίση τεράστιων διαστάσεων ώστε η Ευρώπη να, να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί. Ωστόσο χάθηκε μια ευκαιρία εν μέρη για να ενισχυθούν τα κοινά θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Διότι αφενός αυτές οι νέες αρχές επιτήρησης εποπτείας έχουν ένα πεδίο αρμοδιοτήτων περιορισμένο σε σχέση με παρόμοιες αρχές κρατών μελών. Και είναι κρίμα επιπλέον ότι δεν προχωρήσαμε σε μια αντίστοιχη ενσωμάτωση και ένταξη όπως εκείνη που δημιουργήθηκε σε σχέση με το κεντρικό σύστημα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Προχωρήσαμε, προοδεύσαμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την να ανεβαίνουμε το βουνό, την αναρρίχηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη, τους ε, μεμονωμένους αγωγητές. Ο κύριος Γκοζές, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, φυσικά συμφωνώ για να συγχάρω. Να συγχαρώ και εγώ στην εξαιρετική αυτή δουλειά, συνεργασία και με το Κοινοβούλιο και να υπενθυμίσω τη θέληση του Κοινοβουλίου. Αυτή η επιτήρηση δεν θα είχε ευρωπαϊκό χαρακτήρα εάν δεν υπήρχε το Κοινοβούλιο όσον αφορά το ΕΚΟΦΗΝ, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι θα ήθελα πριν το τέλος αυτής της περίοδου, ίσως πριν το τέλος αυτού του μήνα, να βρεθεί μια λύση για το θέμα που σας απασχολεί και εσάς και που είναι σοβαρό και που είπατε ότι δεν θα ασχοληθείτε επιματέω. Να βρεθεί μια ικανοποιητική οικονομική λύση για το θέμα του private equity με τη βοήθεια της Βελγικής Προεδρίας. Έχουμε τη συνήθεια εικόνα του Επιτρόπου σε αυτό το πλαίσιο να προσφέρει τα τους, τα, λιθαράκια που θα οικοδομήσουν έξυπνους θεσμούς. Δεν είναι θέμα ρυθμίσης, είναι θέμα αποτελεσματικότητας ενός κανονισμού που σκοπό έχει να περιορίσει όσο αυτό γίνεται τους ενδογενείς κινδύνους του χρηματοπιστωτικού ε, ε, συστήματος. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον David Wright που δυστυχώς μας φεύγει. Ελπίζουμε ε, με όλη τη δουλειά που έκανε για να βοηθήσει το κοινοβούλιο μας ε, για να κάνει αυτό το έργο να τον βρούμε κι αλλού στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ο κύριος Σάντσες Πεσέντο, δυόμιση λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μπαρνέ, Επίτρο, ε, Υπουργέ Ρέντε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω το συμβιβασμό που επετέφθη για να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και με επιτυχία το πακέτο για την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Αυτό ήταν ένα παλιό αίτημα για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ένα απαραίτητο μέσο για να προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση την χρηματοοικονομική κάνοντας πιο αποτελεσματική την νομισματική πολιτική και βελτιώνοντας τον ανταγωνισμό. Ήταν κάτι που εκκρεμούσε ώστε να θέσουμε όρια στις ε, αλόγιστες πράξεις, να ελέγξουμε τι πράξει και με μια διεθνή επιτήρηση. Η σημερινή κρίση επικύρωσε την επάρκειε ε, των αγορών ε, και σε σχέση και με τα εθνικά επίπεδα. Πρέπει να διορθώσουμε, να επανορθώσουμε τα σφάλματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί. Στη δική μας περίπτωση η εποπτεία έχει προτεραιότητα, διότι αν η ευρωπαϊκή ρύθμιση ήταν ελληματική, η εποπτεία ήταν ανύπαρκτη. Η ευρωπαϊκή εποπτεία δημιουργεί τα θεμέλια για μια πλήρη μεταρρύθμιση σε βάθος και αξιόπιστη αυτή η πρώτη θα έλεγα διεθνική εμπειρία είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός για μια διεθνή εποπτεία εργάστηκε ενωμένο το Ευρωκοινοβούλιο ώστε αυτό το πακέτο μέτρων να έχει τη σωστή κατεύθυνση, να είναι πιο ισόρροπο λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων, την προστασία των καταναλωτών, των φορολογουμένων και να είμαστε πιο λογικοί στην αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων, να δρούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να αντιμετωπίζουμε τα τοξικά προϊόντα και μεγαλύτερη αηφορία λόγω της βελτίωσης στον ανταγωνισμό, ρυθμίζοντας τα, τα κόστη και έτσι έχοντας ένα σύστημα διαχείρισης διαχείριση κρίσεων που θα βασιζόμαστε για αυτή τη διαχείριση στις αναγκαίε νέε αρχές. Η δρομολόγηση αυτή των αρχών ε, με το μειακό χαρακτήρα, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, θέτοντα κανόνες για τη λειτουργία τους, όλα αυτά βελτιώνουν και αυξάνουν τον ανταγωνισμό και βελτιώνουν και δίνουν δυνατότητες συνεργασίας. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα μέσα σε προθεσμία να ολοκληρωθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2012 αυτό το μέτρο και να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε πλήρια αρμονία. Χαιρετίζω και συγχαίρω εκείνου που κατέστησαν εφικτό να προχωρήσει αυτό το πακέτο. Σήμερα ντρέπουμε του πρώτου καρπού. Αυτό ο συμβιβασμό χαρακτηρίζει τη διαχωριστική γραμμή για αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Διότι η δημοκρατία πρέπει να νομοθετεί και να επιτηρεί. Να διασφαλίζει ότι θα συμμορφώνονται όλοι προ του νόμου. Γι' αυτό όσοι θέλουμε καλύτερα χρηματοοικονομικά πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική δημοκρατικότητα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γκουλάρ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, πολλά υπόθηκαν. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία, είναι ικανοποιητική. Ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα ένα μάθημα να αντλήσω για το μέλλον. Η συναπόφαση δεν μπορεί να είναι όπως έκανε τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΚΟΦΗΝ με, να πετυχαίνουν ομοφωνία στο Συμβούλιο και να έρθουν στο Κοινοβούλιο και να είναι κρίμα, κρίμα, κάντε το γρήγορα γιατί εμείς συμφωνήσαμε. Η, κύριε Υπουργέ, ε, ευχαριστούμε τη Βελική Προεδρία γιατί παλέψτε λίγο περισσότερο για το σημείο αυτό. Να σας πω ωστόσο το εξή Για την οικονομική διακυβέρνηση, όπως και για την εποπτεία, πρέπει να δουλέψουμε ομαδικά. Άρα, ή δυνατόν κύριε Ρέντες, περάστε ένα μικρό μήνυμα στους συναδέλφους σας και εσείς κύριε Μπαρνιέ στο ΕΚΟΦΗΝ. Θέλουμε να μετέχουμε εξ αρχής πλήρως και να παίζουμε το ρόλο μας στην συναπόφαση. Μην έρχεστε με ένα έτοιμο κείμενο από το Συμβούλιο ή την Task Force. Και μετά εξηγήστε στον κύριο Βαν Ρόμποϊ ότι θα θέλαμε να τον βλέπουμε στην Οικονομική Επιτροπή όπως το ζητήσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέρμπερ. ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, όχι μόνο για το ευρωπαϊκό όργανα, αλλά και για τον Ευρωπαίο πολίτη. Μετά τη Lehman Brothers πέρασαν δύο χρόνια και καταφέραμε τελικά να βρούμε μία λύση που μπορεί να μην λύνει όλα τα προβλήματα, θα συμβάλλει ωστόσο στην αποφυγή των υπερβολών ε, των τραπεζών στην Ευρώπη. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Προεδρία του Συμβουλίου, τη Βελική Προεδρία, και να υπογραμμίσω αυτά που είπε η κυρία Γκουλάρ προηγουμένως. Στο ξεκίνημα τα πράγματα ήταν εύκολα, θεωρούσαμε. Πήρε ομόφωνα απόφαση το Συμβούλιο, δεν λύθηκε το πρόβλημα ωστόσο και νομίζω ότι το καλό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ξεπέρασε τις κομματικές αντιπαραθέσεις για να βρει μια λύση που στέκει και που θα επιτρέψει να αποκτήσουμε στέρεες δομές εποπτείας και κατά συνέπεια θα αποτελέσουν εργαλείο που σε μια στιγμή κρίσης θα επιτρέψουν την προστασία και τη σταθεροποίηση του κλάδου του οικονομικού κλάδου. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Ρέντερς, κάνατε καλή δουλειά, δείξατε ε, πάθος και να ευχαριστήσω επίσης και την Επιτροπή που διεξήγαγε ένα δίκαιο, σωστό διάλογο επιτρέποντας να υπάρξει προσέγγιση των θέσεων όλων των πλευρών. Ευχαριστώ εκ νέου για την δουλειά σας αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φτρεμόσε, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτομάτως την επόμενη πενταετία θα γίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού συστημικού κινδύνου. Αυτό είναι σοβαρό γιατί σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμπλέκεται στην ευρωπαϊκή επιτήρηση μαζί με άλλους θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Ο κύριος Τρισέ δηλαδή, ο οποίος είναι υπόλογος στο κοινοβούλιο αυτό, θα πρέπει να απαντά επίσης και σε ερωτήματα ε, που αφορούν την δημοσιονομική επιτήρηση και όχι μόνο ερωτήματα που έχουν σχέση με την σταθερότητα των τιμών. Με την μεταρρύθμιση αυτή, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέτει σε κίνδυνο την φήμη του και την αξιοπιστία του για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Το να κάνουμε λοιπόν τη δουλειά μας όπως συνήθως θα είναι πιο δύσκολο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προκάλεσαν αυτή την κρίση και ε, θα ε, ευχαριστήσει αυτό τους, τις μελλοντικές γενναίες των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λούλιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτούς που χαίρονται εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, ε, το χρηματοπιστωτικό αυτό πακέτο εποπτείας. Το, αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό, όχι μόνο γιατί το Συμβούλιο ε, αντιστάθηκε στους εκπροσώπους του κράτους, ε, αλλά επειδή έχει βαρύτατο νόημα, έπρεπε να δώσει μια ευρωπαϊκότερη διάσταση στο πακέτο, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του. Η κυρία Γκουλάρ και εγώ ως σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μας δώσαμε μεγάλες μάχη ώστε ο πρόεδρος Κεντρική Κεντρικής Τράπεζας εξοφίσιο να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Το κάναμε επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη, σημασία του θέματος. Σε ένα χώρο που θα παραμείνει κατακαιρματισμένο μεταξύ των εθνικών αρχών χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό όργανο που θα είναι ισχυρό, θα έχει αρμοδιότητες και θα νομιμοποιείται χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό θα το καταλάβουν πιθανώς ακόμα και οι Βρετανοί. Ε, θα, χάρη στην, ε, το γόητρό του και στην εξουσία που έχει θα μπορέσει να, επιβάλλει, να επιβληθεί από αυτό το όργανο απέναντι στους διάφορους συνομιλητές του, κυρίως τους υπουργούς. Δεν υπάρχει υπερβολική εξουσία που πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε. Είναι η υπερβολική αδυναμία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, ε, πρέπει όλες οι αρχές που θα αποφασίσουμε σήμερα να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους. Δεν έχουμε ακόμα κερδίσει. Πρέπει για μία ακόμα φορά να παραδεχτούμε ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε αλλά τελικά σήμερα σήμερα ε, δημιουργούμε τις ενδιαφέρουσες βάσεις ενός μοντέλου που θα κληθούμε να αξιολογήσουμε τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τη διαδικασία του Catch the Eye. Δυστυχώς το λόγο θα δώσουμε μόνο σε πέντε συναδέλφους. Ο κύριος Παλώνε, ένα λεπτό συγγνώμη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε πεπισμένοι ότι στην παγκόσμια αγορά κανένας, κανένας ε, ε κανένα προϊόν δεν μπορεί να αποφύγει την ε, σωστή ρύθμιση και έλεγχο. Η πρόσφατη κλίση έδειξε την αναγκαιότητα να, να λαμβάνονται αποφάσεις 48 ώρες, άρα χρειάζονται κοινοί κανόνες. Οι too big to fail πρέπει να εποπτεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κόστος δεν πρέπει να το υφίστε το πολίτης. Κατά συνέπεια χρειάζεται διαφάνεια, ευθύνη και έλεγχος επικροτώ την συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσα σε συμφωνία στην οποία το Κοινοβούλιο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητων αρχών με ε, δυνατότητες επιβολής κυρώσεων και επέμβασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνο με την δημιουργία ε, δομών που δεν μπορούν να φόρουν ότι οι φόροι και στις συναλλαγές δεν μπορεί να είναι ε, μία λύση μόνο και Πιστεύω ότι χρειάζεται, κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό διότι δεν έχουμε ενιαίο τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Κούτας, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω το γεγονός ότι κινούμεθα από μια κατακαιρματισμένη δομή επιτήρησης και εποπτείας που χαρακτηριζόταν από αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο σε μια κοινή εποπτεία ευρωπαϊκού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή φωνή. Θα μπορέσει μακροοικονομικά να αναλάβει δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή της για να αποφύγουμε μια μελλοντική χρηματοοικονομική κρίση. Τα κράτη-μέλη αγνόησαν, αγνόησαν την πρόταση των Ευρωβουλευτών να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων. Θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε όμως το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι μία από τις πηγές συστημικών κινδύνων. Τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμά τους να διαφωνήσουν και να έχουν δικαίωμα ένσταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή. Όμως η περίοδος των μικρών βημάτων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Χρειαζόμαστε πλήρη πολιτική εμπλοκή για να προχωρήσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Γιάτεν Μάκη. Παρακαλώ. Η κυρία Γιάτεν Μάκη, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο ευρωπαϊκού χαρακτήρα λύσεις και χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό από πλευρά εθνικού επίπεδου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματήσει εδώ η δουλειά. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να το ξαναδούμε. Πρέπει να περιορίσουμε τους κινδύνους ε, όσον αφορά τις τραπεζικές δραστηριότητες που ξεπερνούν το 70%. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εποπτεία, περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία που είναι, θα είναι προς το κοινό συμφέρον και θα διασφαλίζει αυτό το κοινό συμφέρον. Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε μια σε μέγιστο επίπεδο θα έλεγα συμφωνία σε σχέση με τις αρχές. Δεν είναι βέβαια ιδανική διότι κάποιες από τις τραπεζικές δραστηριότητες παραμένουν ακόμα στα χέρια και στα συμφέροντα των κρατών μελών που είναι ας το πω έτσι διαχωρισμένα μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Grazie. Ο κύριος Μπρόντς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κόσμος θεωρεί ότι η κρίση είναι καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τι κρίσει ω ευκαιρίε για να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες, πάντα ει βάρο των εθνικών κυβερνήσεων. Τα κράτη-μέλη χάνουν την κυριαρχία τους στα χρηματοοικονομικά του συστήματα. Είναι γεγονό ότι η κρίση στη Βρετανία αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά κακό τρόπο. Αλλά αυτό ήταν διότι οι διάφορες ε, διαδοχικές βρετανικέ κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να ελέγξουν τις δραστηριότητε του private, ε, του private banking. Οι τράπεζε κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα μόνες τους. Δημιουργούν το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο τμήμα της πίστοση ε, που παραμένουν στα χέρια των ιδιωτών και αυτό είναι καλύτερο. Ευχαριστώ τελευταίος αυτό το πλαίσιο, Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι ο συμβιβασμός είναι ένα ορόσημο στην περαιτέρω εξέλιξη συνολικά της ευρωπαϊκής εποπτείας και σε σχέση και με το θετικό πνεύμα με το οποίο συνεργάστηκε η Προεδρία του Συμβουλίου και που ε, χάρη στις διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τα κράτη-μέλη επετέφθη αυτός ο ε, συμβιβασμός. Έχουμε δημιουργήσει τώρα φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς που μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά όταν χρειαστεί. Και έτσι σε σχέση με την αρμοδιότητα θα είναι δεσμευτική η τοποθέτηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και όχι πλέον των εθνικών εποπτικών αρχών. Χρειάζονται λοιπόν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό σύστημα θα είναι υπό την εποπτεία του ε, Προέδρου που ε, θα ε, μπορεί έτσι να είναι αποτελεσματικό. Χαίρομαι και ευχάζω τι ευχαριστίες μου από πλευρά τη κομματική μου ομάδα για την καλή αυτή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπο κύριος Μπαρνιέ. Παρακαλώ του συναδέλφου, να μην μιλάνε. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθώς ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, τους υπευθύνους των ομάδων, όπως και τα μέλη του Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο. Ομόφωνα σχεδόν για να στηρίξουν το συμβιβασμό αυτό και την συμφωνία επιβεβαιώνω ότι αυτές οι νέες ευρωπαϊκές αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων δεν θα υποκαταστήσουν τις εθνικές αρχές εποπτείας αλλά θα στηριχθούν σε αυτές θα τις κάνουν να συνεργαστούν καλύτερα. Η πρόεδρος φωνάζει «Παρακαλώ συνάδελφοι κάντε ησυχία». Θα μπορέσουν λοιπόν να δικτυώσουν τις αρχές αυτές μεταξύ τους για να αλληλοσυμπληρώνονται οι αρμοδιότητες και οι ειδικέ γνώσεις ώστε να υπάρχει μια καλή ευρωπαϊκή απόκριση όποτε αυτό χρειάζεται απέναντι σε κινδύνους ευρωπαϊκούς ή και μεγαλύτερους στις χρηματοοικονομικές αγορές που όπως σας είπα είναι κυρίως υπερεθνικές. Χάρη σε εσά λοιπόν και χάρη στο Συμβούλιο θα υπάρξει αυτό. Πρέπει να συμπληρωθεί σιγά σιγά. Θα πρέπει το, το, ε, το σύστημα πληρωμών, το ΣΕΠΑ, από τον Οκτώβριο, ο κανονισμός για τα ίδια κεφάλαια, η μεταρρύθμιση της ε, οδηγίας για τις αγορές, ε, για τις χρηματοοικονομικές αγορές, για τους καταθέτες, τους, τις, τους οργανισμούς αξιολόγησης και μια σειρά από άλλα είναι νομοθετήματα έχουμε ακόμα να προχωρήσουμε θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα ώστε στο τέλος, εν κατακλείδη, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι βουλευτές, και όπως έχουμε ως οδικό χάρτη από τις συνεδρίες των G8, κανένας παράγων, κανένα προϊόν, καμία αγορά, καμία περιοχή να μένει εκτός αυτής της ευφυούς και αποτελεσματικής νομοθεσίας. Στόχος μας, φιλοδοξία μας είναι από κοινού στο τέλος αυτού του σύντομου δρόμου, γιατί περιμένουν δικαίως οι πολίτες πολλά από μας να έχουμε οικοδομήσει από κοινού κυρίες και κύριοι και όχι με καθυστέρηση το καλύτερο παγκόσμιο σύστημα ρύθμισης και εποπτείας. Η Ευρώπη θα πρέπει να θέσει στόχο της να οικοδομήσει ένα δικό της μοντέλο ρύθμισης και εποπτείας, το καλύτερο στον κόσμο. Αυτό είναι ο στόχος μας, η φιλοδοξία μας υπέρ των καταναλωτών και βεβαίως του ίδιου του χρηματοοικονομικού κλάδου. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο Υπουργός κ. Ζέντερς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλου όσοι έλαβαν το λόγο, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων υποστήριξαν ε, τα κείμενα που έχετε ενώπιόν σα προ ψήφιση. Δείχνει, νομίζω, το ενδιαφέρον που πάρα πολλοί βουλευτέ έδειξαν για το ζήτημα και για την χρηματοοικονομική εποπτεία εν γέννη. Να σα πω καταρχά ότι όπω πολλοί υπενθύμησαν είναι αυτό το πρώτο πραγματικό μάθημα που λάβαμε από τη χρηματοοικονομική κρίση. Συζητήσαμε μακρόν το κείμενο, η δημιουργία ωστόσο αυτής της νέας εποπτικής δομής, η δημιουργία του οργανισμού ε, ελέγχου του συστημικού κινδύνου είναι το πρώτο μάθημα που παίρνουμε στην Ευρώπη για την κρίση, από την κρίση. Δεύτερο στοιχείο. Πρόκειται για ένα ξεκίνημα. Ο κ. Μπαρνιέ το υπενθύμησε. Θα θεσπίσουμε μια σειρά άλλων δομών και στοιχείων στη διαδικασία αυτή. Η ρυθμιστική αντιμετώπιση θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο την συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η Βελγική Προεδρία είναι από πλευρά τη απόλυτα αποφασισμένη να συνεχίσει στην ίδια πορεία. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην οδηγία για τα ε, επενδυτικά τα ταμεία επενδύσεων. Θα γίνουν οι συζητήσεις για τις οργανισμούς ε, αξιολόγησης. Ήδη έχουμε προτείνει και έχει συμφωνηθεί στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ να είναι παρούσα και η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κυρίας Μπόλς για να ενημερωθεί για το πώς προχωρούν οι εργασίες μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσει ότι ξέρω ότι ακολουθούν ψηφοφορίες. Να σας πω ωστόσο ότι ελπίζω πως θα μπορέσουμε να δούμε μια πραγματικά όπως πολλοί ανέφεραν ιστορική ψηφοφορία και ελπίζω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αποφασιστικότητα και άλλα σημαντικά κείμενα που θα σας υποβληθούν εκ νέου. Ευχαριστώ εκ νέου όλους όσοι τους τελευταίους μήνες επέτρεψαν να προχωρήσουν τα ζητήματα αυτά που επαναλαμβάνω αποτελούν το πρώτο σημαντικό μάθημα που λάβαμε από τη χρηματοοικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Περαιούται η συζήτηση. Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα. Βλέπω ότι εν μέσω ημών βρίσκεται μια νεότατη συνάδελφος, η μικρή Βιτόρια, κόρη της κυρίας Ροντζούλη. Να συγχαρώ και τη συνάδελφο και την κόρη της συναδέλφου. Να τη συγχαρώ νομίζω εξ ονόματος όλων των μελών του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Σύντομα, κύριε συνάδελφε. Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ. Είμαι εδώ συμβολικά με την κόρη μου Βιτόρια και θέλω να σκεφτώ όλες εκείνες τις γυναίκες που για λόγους εργασίας δεν μπορούν να συμφιλιώσουν την ε, εγκυμοσύνη και την επαγγελματική ζωή με την οικογένεια. Νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να τους αφήσουμε να παίξουν καλύτερα το ρόλο της μητέρας και ζητώ μια καλύτερη παρέμβαση της, ε, των Ευρωπαϊκών Οργάνων και του Κοινοβουλίου για να μην μπορεί ε, μια γυναίκα ποτέ να ξαναβρεθεί στο δύσκολο αυτό σταυροδρόμι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Συγχαρητήρια εκ νέου ενστερνιζόμαστε την έκκληση που απευθύνεται με τόσο θερμό τρόπο. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες.